Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Καμία αντίρρηση. Εγκρίνονται. Le deuxième point à l'ordre du jour, l'adaptation des procès-verbaux des réunions précédentes. Έγκριση των πρακτικών του Μαρτίου και του, της 5ης Απριλίου του 2011 το έχετε λάβει αν έχετε παρατηρήσεις δυστυχώς η διερμηνία γίνεται με μεγάλη δυσκολία λόγω ναι. ενός μικροφωνισμού εγκρίνονται και τα πρακτικά δεν έχουμε λάβει καμία ερώτηση προς την Κομισιόν Όσον αφορά στις ανακοινώσεις, ε, δεν έχω καμία ανακοίνωση. Η Επιτροπή έχει κάτι να μας πει. Α, επιτέλους. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους. Μπορεί, αυτά είναι οι αργίες, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένη, δεν έχουμε την πληροφορία. Δεν έχουμε το περιοδικό μαζί. Θα αλλάξω μικρόφωνο, λέει η σοφά η πρόεδρος. Αυτό το μικρόφωνο είναι καλύτερα, ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό το μικρόφωνο θα κρατήσω, λοιπόν. Έξι εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012. Η Επιτροπή μας ε, προετοιμάζει γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον Τρίλογο σχετικά με τον προϋπολογισμό 2012. Ο κύριος Γκέρενς είναι ο εισηγητής μας και θα του δώσω το λόγο ευθύ αμέσω. Κύριε Γκέρενς για τη γνωμοδότησή σας, για τον τρίλογο. Μπορείτε να μου δώσετε πέντε λεπτά για να μπορέσω κι εγώ λίγο να συγκεντρωθώ για το θέμα και να προχωρήσετε με κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι το επόμενο σημείο είναι επίσης δικό σας. Είστε εσείς ε, η βεντέτα της ιστορίας. Θέλετε το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης Μα η ομάδα σας τα είχε καθορίσει αυτά. Τότε πάμε στο επόμενο, πάμε στο σημείο 8. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γκορ. Θα κρατήσει μία ώρα, κύριε Γκέρενς. Έχετε λοιπόν μία ώρα για να προετοιμαστείτε. Όπως όλοι σας γνωρίζετε, η τέταρτη διάσκεψη του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη από τις 9 έως τις 13 Μαΐου. Στόχος ε, της διάσκεψης είναι να αξιολογήσει τα δεκαετή σχέδια, τον απολογισμό του δεκαετού σχεδίου δράσης ε, που εγκρίθηκε στις ε, Βρυξέλλες το 2001 και το τι θα γίνει για την επόμενη δεκαετία. Στις 3 Μαρτίου, στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με τον κύριο Ντιάρα, τον ε, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΙΕ αρμόδιο για την Αφρική και είπα του αρμοστή για τις ΛΑΧ, μας ανέφερε σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης, την προσαρμογή του προγράμματος των Βρυξελών και του ορισμού των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη των ΛΑΧ. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εγώ υποδέχομαι τον κύριο Σάρλ Γκοχ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την Αφρική στην UNCTAD για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και ασχολείται με τις ΛΑΧ. Εδώ και 10 χρόνια ασχολείται με το θέμα. Και πριν του δώσω το λόγο θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω το έργο της UNCTAD η οποία κατάφερε να δημιουργήσει την κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των ΛΑΧ και τις βοηθάει σε διεθνές επίπεδο. Κύριε Γκόρ, σας δίνω το λόγο για 20 λεπτά. Um, thank you. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα ευγενικά σας λόγια προς την UNCTAD και τη δουλειά μας. Με μεγάλη ευχαρίστηση προσήλθα σήμερα εδώ και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικότερα μηνύματα ή συμπεράσματα της τελευταίας μας έκθεσης που λεγόταν προς μια νέα διεθνή αρχιτεκτονική ανάπτυξη για τη ΣΛΑΧ. Η δε παρουσίασή μου που δεν βλέπουν οι διερμηνείς θα αφορά τρία βασικά θέματα. Το ένα είναι πώς τα κατάφεραν οι ΛΑΧ κατά την περίοδο 2000 με 2010. Δεύτερο ερώτημα. Πώς προχώρησε η σφαιρική συμφωνία για εταιρική σχέση και τρίτον τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί αυτή η λεγόμενη global partnership. Τώρα, αν δούμε Πώς τα κατάφεραν οι ΛΑΧ την, την περασμένη δεκαετία, όπως και οι υπόλοιπες χώρες πέρασαν από ένα κύκλο ανάπτυξης και έναν κύκλο ύφεσης και μέχρι την έκρηξη της δημοσιονομικής ή χρηματοπιστωτικής κρίσης του 8 ευημερούσαν. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ τους ήταν υψηλότερος από ό,τι άλλων αναπτυσσομένων χωρών και υψηλότερος από των ανεπτυγμένων 8 περίπου, όχι, ο ρυθμός αυτός ανάπτυξης ανταποκρινόταν πάνω κάτω στους στόχους που είχαν τεθεί που ήταν πολύ ψηλότερος από τη δεκαετία του 90 και του 80. Στους κύκλους της ύφεση η ΛΑΧ αντιστάθηκαν καλά και κατ' εμάς η αντίσταση αυτή παρόλα αυτά είναι δεν είναι αληθινή διότι οφείλεται στο ότι οι τιμές των εμπορευμάτων διατηρήθηκαν απλώς. Η ανάπτυξη δηλαδή δεν ήταν τόσο καλή όσο φαινόταν. Παρά το σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, οι ΛΑΧ διαχωρίστηκαν από τις υπόλοιπες χώρες γιατί είχαν πολύ χαμηλή δυνατότητα παραγωγής και η μείωση της ανέχειας έγινε με πολύ χαμηλό ρυθμό. Το βασικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι υπήρξε μαζική ανάπτυξη αλλά πολύ βραδία καταπολέμηση της ανέχειας. Πώς γίνεται αυτό. Βλέπουμε, παρατηρήσαμε ότι είναι πολύ χαμηλές οι δυνατότητες παραγωγικότητας στις χώρες αυτές. Η γεωργία, η παραγωγικότητα της γεωργίας αναπτύσσεται με πάρα πολύ βραδύ ρυθμό και αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες οι χώρες αυτές για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους εκτός της γεωργίας. Ε, Επίσης πολύ ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται οι εισαγωγές τροφίμων και φτάνουν τα 24 δισεκατομμύρια έφτασαν το 2008. Η στατιστική για την ανέχεια δείχνει ότι, οι στατιστικές, ότι η κατάσταση στις ΛΑΧ χαρακτηρίζεται από μαζική ανέχεια. 50% του πληθυσμού ζουν με κάτω από ένα δολάριο την ημέρα. 421 εκατομμύρια ανθρώπους αφορά αυτό και θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα τρίτο περίπου του συνολικού αριθμού των πτωχοτέρων παγκοσμίω. Um, that shows um, the εδώ βλέπετε ότι ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τον στόχο. Υπήρξε μία καμπή το 1994, δηλαδή, δηλαδή μέχρι τότε αυξανόταν οι δείκτες και μετά άρχισαν να πέφτουν αργά αλλά σταθερά και η πτώση αυτή επιταχύνθηκε μετά. Η ανέχεια δηλαδή μειώνεται πάρα πολύ αργά και πολύ βραδύτερα από ό,τι προέβλεπαν οι στόχοι, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας, η ΑΣΧ. και παρά την μείωση αυτήν μπορεί να αυξάνεται και ο αριθμός των πτωχών όσων ζουν δηλαδή με κάτω από ένα δολάριο την ημέρα. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 100% το 2007 σε σύγκριση με το 1980. Η πρόοδος των ΑΣΧ στα ΛΑΧ δείχνει ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος. Η πρόοδος δηλαδή αυτή είναι πολύ ευραδία και αυτή. Αφ, γρήγορη ανάπτυξη αλλά βραδία πολέμηση της ανέχειας. Πολύ σημαντικό αυτό το συμπέρασμα. Και εδώ βλέπετε ότι η κύρια αναπτυξιακή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ΛΑΧ είναι πώς να δημιουργήσουν παραγωγικές θέσεις απασχόλησης και εισοδήματα για το εργατικό δυναμικό που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Μόνον εάν δημιουργηθούν παραγωγικές θέσεις απασχόλησης και εισοδήματα. Ποια είναι η κλίμακα της πρόκλησης λοιπόν. Από το Μαλί και τη Μαδαγασκάρη βλέπουμε ότι οι αριθμοί δείχνουν ότι η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, η δημογραφική ανάπτυξη δηλαδή, ο αριθμός των ανθρώπων μεταξύ 50 και 60 ετών αυξάνεται. Στο Μαλί το 2005 δημιουργήθηκαν 271.800 θέσεις εργασίας, αλλά ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κάθε χρόνο αυξάνεται μέχρι να φτάσει στην ακμή του στο, στις 447.000. Αν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε την ανεργία στο Μαλί, την ανέχεια μάλλον, θα πρέπει να αλλάξει ο ρυθμός αυτός που αυξάνεται κάθε χρόνο. Στο Μαλί προβλέπεται το 2045 να καμφθεί η τάση αυτή. Βλέπετε εδώ ποιες είναι οι προκλήσεις, οι αναπτυξιακές προκλήσεις. της ΛΑΧ από το 2005 μέχρι το 2015 αν δεν αναπτυχθούν αυτά, αυτές οι παραγωγικές θέσεις εργασίας και εισοδήματα θα αυξηθεί η ανέχεια. Δεύτερον, αυξάνεται η μετανάστευση από τις χώρες αυτές. Άρα, αυτή είναι η πρόκληση, αυτό είναι το κύριο θέμα. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε μια πρόσθετη διάσταση του προβλήματος για την επόμενη δεκαετία. Αν ήμασταν εδώ το 1980 θα βλέπαμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που μπαίνουν στην εργασία το έπραταν στην γεωργία. Και αυξάνονταν και ο αριθμός των καλλιεργησίμων γεών. Αλλά η τάση αυτή απορρόφησης των εργαζομένων από την Γεωργία άρχισε να μειώνεται διότι άλλαξε η πυκνότητα του πληθυσμού και φτάσαμε σε όρια γεωκτησίας. Είναι δηλαδή άνθρωποι τόσο πτωχοί που δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα μέσα και πόρους για να αποκτήσουν άλλα χωράφια. Σημειώνεται λοιπόν μια αλλαγή. Όλο και περισσότεροι ψάχνουν εργασία εκτός της γεωργίας που παραμένει όμως ο κύριος πόρος εισοδημάτων στις χώρες αυτές αλλά όλο και περισσότεροι νέοι ψάχνουν δουλειά εκτός γεωργίας. Η γεωργία, οι γεωργικές δραστηριότητες αυξάνονται πολύ πολύ αργά και είναι σχεδόν αδύνατον να δημιουργηθούν παραγωγικές θέσεις και εισοδήματα εκτός γεωργίας, στη βιομηχανία ή στις υπηρεσίες δηλαδή. Σημειώνεται μια αλλαγή όπου, σύμφωνα με την οποία μάλλον, η περισσότερη πτωχή αυτή τη στιγμή δεν είναι πια στη γεωργία αλλά εκτός αυτής. Εδώ υπάρχει, βλέπετε και μια γελιογραφία που δείχνει την παγκόσμια κατάσταση. Υπάρχουν κλιματολογικές αλλαγές που είναι ήδη πραγματικότητα στις χώρες αυτές και υπάρχουν και νέες χρηματοπιστωτικές προκλήσεις καθώς και μεγαλύτερη πτητικότητα των τιμών. Υπάρχει λοιπόν η πρόκληση της ανεργίας, οι κλιματολογικές αλλαγές. Οι ΛΑΧ θέλησαν να ανοίξουν την οικονομία τους και να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες παγκοσμίω και τέλος υπάρχει και η πρόκληση της διακυβέρνησης ή της διαχείρισης. Εδώ τονίζω ότι απαραίτητος θα υπάρξει και τέτοια κρίση, δηλαδή διαχείρισης. Είναι απλώς θέμα χρηματοπιστωτικών πόρων. Οι ΛΑΧ, όπως δείχνω εδώ, έχουν μέσω ΑΕΠ κατά κεφαλήν 1 δολάριο λεπτά ενώ η κατανάλωση, η ημερήσια κατανάλωση ανά νοικοκυριό είναι ένα δολάριο κόμμα 14. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες αυτές κατά μέσο όρο έχουν 45 λεπτά αναπρόσωπο και αναημέρα διαθέσιμα για επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. 45 λεπτά δαπανούν 20 από αυτά την ημέρα για την διακυβέρνησή τους. Ο αριθμός κάτω-κάτω δείχνει τι ισχύει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι λάθος η διαφάνεια. Όπου προβλέπονται 20 δολάρια ανά άτομο ανά μέρα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί προσπαθούν να καταφέρουν με 20 λεπτά την ημέρα. 20 cents και τα χρήματα που διαθέτουν που είναι 45 λεπτά την ημέρα για δημόσια και ιδιωτική επένδυση και για διακυβέρνηση πώς μπορεί μια κυβέρνηση να λειτουργήσει συνάντησα πρόσφατα έναν συνάδελφο που ήταν διπλωματικός στο, Λεπάν, στο Νεπάλ και κέρδιζε ως διπλωματικός 300 δολάρια το μήνα. Έτσι δουλεύουν αυτού του είδους οι κυβερνήσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση, η απασχόληση και η διακυβέρνηση. Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργήσε η εταιρική σχέσης υπήρξε πρόοδος. Το πρόγραμμα δράσης των Βρυξελών που συμφωνήθηκε εδώ μέσα πριν από 10 χρόνια ήταν πολύ αποτελεσματικότερο από ότι τα πρώτα δύο προγράμματα δράσης. Και αυτό θέλω να το δηλώσω, να το τονίσω, πιο αποτελεσματικό. Το πρώτο πρόγραμμα είχε ιδεολογικά προβλήματα, δηλαδή βασιζόταν σε κρατικές επενδύσεις για την ανάπτυξη. Βασικά δηλαδή ήταν άσχετο τελείως. Και οι ΛΑΧ ανέλαβαν την υποχρέωση να κάνουν πλήρη σχεδόν απελευθέρωση των οικονομιών τους, αλλά αυτό έγινε με ασυμμετρικό τρόπο, δηλαδή οι αναπτυξιακοί εταίροι μείωσαν σημαντικά τη βοήθεια που χορηγούσαν. Τσάι παρακαλώ, τσάι. Ενώ στο αναπτυξιακό πρόγραμμα των Βρυξελών ήταν πιο αποτελεσματική η βοήθεια όταν κάναμε την αναθεώρηση ή αξιολόγηση των μέτρων που είχαν εφαρμοστεί για τις ΛΑΧ, διαπιστώσαμε ότι είχαν μάλλον συμβολική σημασία παρά πραγματική και αναπτυξιακή. Το πρόγραμμα δράση των Βρυξελών λοιπόν προβλέπει 156 δράσεις που ανέλαβαν, που υποσχέθηκαν να εφαρμόσουν οι ΛΑΧ Αναλύσαμε 8 όπως ο στόχος του 0,15% ειδικές, ειδικά μέτρα για πρόσβαση στον ΠΟΕ, για την εφαρμογή των συμφωνιών τα πάντα πληνόπλων και από τις αξιολογήσεις αυτές που έγιναν επανειλημμένα είδαμε τα ίδια συμπεράσματα να προκύπτουν ότι τα αναπτυξιακά ωφέλη περιορίζονται λόγω δομικών προβλημάτων στα προγράμματα και λόγω προβλημάτων στην εφαρμογή τους. Για όσο για τη χρηματοδότηση, πολύ λίγα χρήματα διατέθηκαν. Δεν θα επισήλθω σε λεπτομέρειες. Πηδήξτε αυτές τις διαφάνειες μερικές από αυτές. Εμείς πιστεύουμε ότι... Ναι, εδώ, εδώ, εδώ σταματήστε εδώ. Αυτά τα ειδικά μέτρα για τις ΛΑΧ λειτουργήσαν μέσα σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο. Um, agenda. Όπως ε, το πρόγραμμα αναπτυξιακής δράσης HIPEC, και άλλα, αλλά υπήρχαν και αδυναμίες και ελλείψεις που πιστεύουμε ότι δεν βοήθησαν τις ΛΑΧ. Ένα βασικό στοιχείο ήταν ότι δεν υπήρχε διεθνής πολιτική για τα προϊόντα. Για τα προϊόντα. Και επίσης η βοήθεια δόθηκε με περιοριστικό τρόπο, επιβλήθηκε. Άρα πρέπει εδώ να καταλάβουμε ότι τα πράγματα βελτιώνονται μεν αλλά τα συγκεκριμένα μέτρα για τις ΛΑΧ έχουν δώσει μάλλον συμβολικά παρά πραγματικά αποτελέσματα και έχουν σχεδόν ακυρωθεί από την επιβολή χρηματοπιστωτικών προγραμμάτων που δεν επαρκούν. Επομένως τίθεται το επόμενο και σημαντικότερο ερώτημα για όλους μας. Πώς θα βελτιώσουμε τη διεθνή βοήθεια και στήριξη στην επόμενη δεκαετία, τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση της σφαιρικής εταιρικής σχέσης. Αυτό είναι το πρόβλημα και το θέμα. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται κάποιο είδους υποδειγμα... Ε, αλλαγή μοντέλου πράγμα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί πολύ εύκολα, πολύ απλά δηλαδή να δούμε ποιο είναι το απραγματοποιητό δυναμικό των χωρών αυτών και όχι μόνο οι ανθρωπιστικές τους ανάγκες. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν στην αγορά της εργασίας μπορεί να αποτελούν ένα τεράστιο δυναμικό. Και το κλειδί εδώ είναι πώς θα πραγματοποιηθεί, πώς θα υλοποιηθεί το δυναμικό αυτό. Αντί για δημογραφικό βάρος δηλαδή να γίνουν όλα αυτά όφελος για τις χώρες ΛΑΧ. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο πρότυπο, στο μοντέλο. Και η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να είναι απλώς χορήγηση βοήθειας. Χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει εμπόριο, τεχνολογία και επενδύσεις και όχι μόνο βοήθεια. Και αυτή η ευρύτερη προσέγγιση πρέπει να δίνει τον κύριο λόγο στις ΛΑΧ και να τονίζει τη βελτίωση των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων Έπειτα, η προσέγγιση βοήθεια συν aid plus δηλαδή απαιτεί συνεργασία με τις ίδιες τις χώρες λάχη, όχι μόνο με τον διεθνή παράγοντα. Και τέλος χρειάζεται αναπτυξιακή συνεργασία νότου-νότου και όχι μόνο βορρά-νότου. Αυτό όμως χωρίς βουρλομανδίες. Αυτά είναι ορισμένα από τα γενικά που διατυπώνουμε στο έγγραφο που ονομάζεται Νέα Αναπτυξιακή Αρχιτεκτονική για τη ΛΑΧ και που βασίζεται στις αρχές που προσπάθησα να σας περιγράψω και σε ορισμένους πυλώνες όπως γράφει εδώ. Έχουμε φανταστεί τι θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, αλλά για να καταλήξω τώρα θα ήθελα να αναφέρω μόνο έναν, μία ιδέα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η βοήθεια. Γιατί μεγάλο τμήμα της αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε κοινωνικούς τομείς και όχι πια σε παραγωγικούς. Γι' αυτό μια μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της παραγωγής για να αυξηθεί και η απασχόληση. Μεγάλο τμήμα είναι παραδοσιακή χρήση της, συνήθις χρήση της βοήθειας, ας πούμε ο εξηλεκτρισμός που είναι ακόμη χαμηλός. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν με, τη συνήθ, με τους τρόπους Παραδείγματο χάρη πώς θα μπορούσε η βοήθεια να χρησιμοποιηθεί για να στηριχθεί η ανάπτυξη των δυνατοτήτων που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες αυτές. υπάρχει εδώ το θέμα των μικροπιστώσεων και των επιχειρήσεων που ε, και της προσπάθειας να έρθουν χρήματα, να δοθούν χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αποτελέσουν τους πρωτοπόρους σε αυτή την προσπάθεια δημιουργίας απασχόλησης. Και εκτός αυτού πρέπει φυσικά να βελτιωθεί και η παραγωγικότητα της γεωργίας και γι' αυτό χρειάζεται και έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό το τονίζω γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρει εσάς ιδιαίτερα αλλά υπάρχουν και άλλε σειρέ μέτρων που τα έχουμε συνοψίσει σε ένα έγγραφο σε ένα φύλλο όπως η πρώιμη συγκομιδή στην Τόχα, μέτρα για τη βελτίωση των πόρων που έχουν οι λάχ, που παίρνουν οι λάχ από τις εξαγωγές τους, μέτρα για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών και τελευταία διαφάνεια εδώ βλέπετε το εξώφυλλο της έκθεσής μας και το βάλαμε για να δείξουμε πόσο ευάλωτες είναι οι χώρες ΛΑΧ, αλλά επίσης γιατί πιστεύουμε ότι η γενικότερη χρηματοπιστωτική κρίση θα μπορούσε να θεωρηθεί θεομηνία ανάλογη με σεισμό που δεν δημιουργεί μόνο, μόνο όμως καταστροφές αλλά δίνει και την ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα και ανοικοδόμηση. Πιστεύουμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή. Η χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει ότι υπάρχει μια ρήξη και αλλαγή και πρέπει να βρούμε νέους τρόπους σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπισης των προβλημάτων και στις ΛΑΧ. Γιατί εκτός από το σύνδρομο too big to fail υπάρχει και το σύνδρομο too small to matter και για τις χώρες αυτές νομίζω ότι τα συμβολικά μέτρα βασίζονται στο φόβο τους ότι μπορεί να μην τους δίνει κανείς καμιά σημασία. Ενώ μέχρι το 2050 θα αριθμούν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Έχουν τεράστιους φυσικούς πόρους, τεράστιο δημιουργικό δυναμικό απραγματοποίητο που σπαταλιέται και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουί Μισελ τώρα το λόγο, ο οποίος είναι και μέλος ε, της Επιτροπής των Σοφών ε, στον ΟΗΟ. Κύριε Μισελ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και ζητώ να με συγχωρήσετε για το αν θα πήγω νωρίτερα γιατί ψηφίζω αλλού. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Σαρλ Γκόρ για την ε, σημαντική του παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία μας ανέφερε, ούτως ώστε να, κινητο... να κινητοποιήσουμε αυτούς που αποφασίζουν παγκοσμίως και που φαίνεται να, είναι, να τσιγκουνεύονται για τις ε, ΛΑΧ. Για την Κωνσταντινούπολη. Είναι μια ομάδα που διορίστηκε από τον κύριο Μπανκιμούν για να προετοιμάσει αυτή τη συνεδρίαση. Αυτό το οποίο πρέπει σίγουρα να πούμε είναι ότι η Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να συνεισφέρει με μια προστιθέμενη αξία έναντι των Βρυξελών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θελήσαμε να περιορίσουμε τις συστάσεις αυτής της ομάδας του ΟΗΕ επί συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες με μια ελάχιστη πολιτική βούληση και ελάχιστα μέσα ε, είναι εφικτές για να μειώσουμε κατά το ίμιση τον αριθμό των ΛΑΧ μέχρι το 2020. Θέλω να αναφέρω τις ε, πρόοδους ε, της τελευταίας δεκαετίας ας πούμε η υγεία, πρόσβαση στο πόσιμο νερό, ε, εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, είχαμε πρόοδους και πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Όχι βέβαια παρκώς, αλλά είχαμε πραγματική πρόοδο. Οι άμεσες επενδύσεις έχουν τέτραπλαστεί, οι υπηρεσίες των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών κατάφεραν να προχωρήσουν με προτιμησιακή μεταχείριση το χρέος μειώθηκε και είχαμε και πολλαπλές προσπάθειες για την μείωση του χρέους. Παρ' όλα αυτά όμως ο απολογισμός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ δεν θέλω να τα ξαναπώ. Ε, το 75% του πληθυσμού των ΛΑΧ ε, ζει με 2 δολάρια την ημέρα, λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, δεν θα φλιαρίσω, θα περιοριστώ για να μην είμαι παναληπτικός για την ε, διακυβέρνηση. Τι εννοούμε εμεί ως διακυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι στη διακυβέρνηση, όλα τα βάζουμε μέσα στη διακυβέρνηση, ακόμη και τον αγώνα για, τις, ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αλλά διακυβέρνηση είναι το τι μπορεί να προσφέρει ένα κράτος προς τους πολίτες του μέσω υπηρεσιών, αντικειμενικών υπηρεσιών, οι οποίες να επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν ε, με αξιοπρέπεια. Πρέπει να βρούμε έναν ορισμό. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορισμένες χώρες αμφισβητούν η γενική δημοσιονομική ε, ενίσχυση ή την τομεακή ενίσχυση. Την αμφισβητούν και αυτό με ανησυχεί σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη. Εγώ είμαι διαυγής και προσπαθώ να είμαι και τίμιος ε, ε, στη σκέψη μου. Αυτή η παγκοσμιοποίηση όπως την είδαμε εμείς ε, τη δεκαετία του 90 ε, που την είδαμε να είναι κλεισμένη, περιχαρακωμένη ε, στα όρια και μόνο της αγοράς αυτό έχει ξεπεραστεί διότι δεν μπορούμε σήμερα να έχουμε μία αξιοπρεπή ε, ε, ε, φιλελευθερωποίηση άμα δεν έχουμε και ένα κράτος που να τη συνοδεύει από δίπλα. Χρειάζεται λοιπόν δημοσιονομική ενίσχυση και τομεακή ενίσχυση προς τα κράτη για να μπορέσουν να οργανώσουν τις υπηρεσίες, διότι χωρίς οργανωμένο και ικανό κράτος είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε ε, να αξιοποιήσουμε σωστά τους φυσικούς πόρους για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα θέμα στη διακυβέρνηση και στην δημοσιονομική βοήθεια. Να ρωτήσω τον κύριο Γκόρ τι σκέφτεται γι' αυτό. Ορισμένε ευρωπαϊκές χώρες δωρητές είναι πολύ επιφυλακτικές και το χρησιμοποιούν αυτό και ως ε, πρόσχημα για να μπορέσουν να μειώσουν τις, ε, ε, την ενίσχυση που δίνουν. Διαπιστώνω επίσης ότι σε ορισμένους κύκλους υπάρχει ψύχωση με την ανάπτυξη. Και εγώ, και εγώ έχω ψύχωση με την ανάπτυξη, αλλά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη χρειάζεται κράτος. Σε ορισμένες χώρες μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη αλλά και αύξηση της φτώχειας. Στη Λατινική Αμερική συνέβη κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Διότι όταν εμείς έχουμε ανάπτυξη αλλά μετά δεν έχουμε μία ανακατανομή αυτού του κέρδους, ε, τότε φυσικά αυξάνει τη φτώχεια. Και σε αυτήν την ομάδα του ΟΗΕ προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα υλοποιούσαμε την ιδέα ενός συμβολέου. Δηλαδή, ένα συμβόλαιο όπου θα είχαμε κριτήρια διακυβέρνησης και όρους ε, διακυβέρνησης συνδεδεμένα με στρατηγικές ε, παραγωγικότητας που θα μας επέτρεπε να δημιουργήσουμε πλούτο. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ανάδυση μιας, ε, μιας μικρομεσαίας τάξης με, τη, με τα μικροδάνεια ή άλλους τρόπους όπως επίσης και στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων που θα πρέπει να διοχετεύονται στην οικονομία να μας πει βέβαια και ο κύριος Γκόρ τι σκέφτεται γι' αυτά. Φυσικά και χρειάζομαι συμμάχους σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία για να πείσω τους Ευρωπαίους ότι δεν ήρθε η ώρα για να εγκαταλείψουμε ε, την ε, τομεακή δημοσιονομική βοήθεια ή τη γενική δημοσιονομική βοήθεια. Ε, σίγουρα πρέπει να έχουμε, ε, να, να, να, να έχουμε, παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας, αλλά γι' αυτό θέλουμε να ε, διαμορφώσουμε αυτό το συμβόλαιο. Αυτά όμως δεν θα τα καταφέρουμε άμα δεν αυξήσουμε την δημόσια βοήθεια, τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να το, το συνδέω με αυτό, με τα αποτελέσματα λέμε. Ορίστε κάθε φορά ο, δώσαμε δισεκατομμύρια και δώσαμε τα δισεκατομμύρια και δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό γιατί, γιατί η κατάσταση παραμένει καταστροφική. Θα ήθελα αυτή την απεσιοδοξία να τη σχετικοποιήσουμε. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε τους ε, τρόπους ε, αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να ενισχύσουμε τα κράτη. Τίθεται το θέμα της συνέχισης της δημοσιονομικής βοήθειας προς τα κράτη. Πρόκειται για πεπιθήσεις που συμμεριζόμαστε, κυρία Πρόεδρε. Ο φόρος των διεθνών χρηματοπιστωτικών πράξεων θα έπρεπε να δημιουργεί να αξιοποιηθεί για την αναπτυξιακή πολιτική. Να πάρουμε περισσότερα ρίσκα. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί φυσικά και οι άλλοι πρέπει να μιλήσουν. Είπαμε, διακυβέρνηση, κράτος, δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια και πώς ε, στην ουσία μπορούμε να ξεκινήσουμε μια πραγματική σχέση συνεργασίας μεταξύ των χωρών αυτών και των δωρητών. Και πρέπει να ενισχύσουμε τον νότο-νότο. Πρέπει να εμβαθύνουμε όλα αυτά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ε, νέα πικιοκρατία στην Αφρική ε, όπου έπικοι θα είναι οι αναδυόμενες ε, δυνάμεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκουερέρο. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Gore, por su presentación hoy en esta comisión. Σας ευχαριστώ. για όλη την προετοιμασία εν ώψη της ε, συνεδρίασης στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από την δαλίστατη ε, τοποθέτηση του κυρίου Μισελ, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία μας είπε, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω μερικά από αυτά που μας είπε. Υπάρχει μία οικονομική φιλολογία η οποία λέει ότι η κρίση που βιώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια είναι η κρίση των ανεπτυγμένων χωρών, είναι η κρίση της φιλελευθεροδυτικής οικονομίας και δεν είναι, πρόκειται για μια κρίση η οποία επηρεάζει τις αναδυόμενες οικονομίες ή τις ΛΑΧ. Αυτό όμως ε, είναι ψέμα. Γιατί. Διότι ορισμένοι δείκτες οικονομικής ανάπτυξης που για πολλές από τις χώρες μας θα ήταν καταπληκτικοί το 3% του ΕΠ είναι ε, ανεπαρκέστατη όχι για να αναπτυχθεί κάποιος παραπάνω, αλλά για να διατηρηθεί το επίπεδο ανάπτυξης πολλών φτωχών χωρών, που για να αναπτυχθούν θα έπρεπε να έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Πήγε μια αντιπροσωπεία αυτής της Επιτροπής ε, στην ε, Βραζιλία και εγώ επήγα κιόλας. Πρόκειται για μια χώρα που αδιαμφισβήτητα έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα στον αγώνα κατά της πείνας, του κοινωνικού αποκλεισμού κλπ. Και μας είπαν ότι αν η ανάπτυξη πήγαινε από το 6% στο 4% πολλές από τις επιτυχίες της Βραζιλίας θα πισωγύριζαν. Αυτές οι χώρες χρειάζονται ένα πολύ ψηλό δίκτυο ανάπτυξης για να μπορέσουν να απορροφήσουν τις ε, νέες ανάγκες για να μπορέσουν να απορροφήσουν και τον νέο πληθυσμό αλλά και να δώσουν δουλειά σε αυτόν τον ενεργό νέο πληθυσμό που όλο ένα αυξάνεται. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις δεν αρκούν οι παραδοσιακές πολιτικές της επίσημης βοή... αναπτυξιακής βοήθειας, την οποία βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε, ε, να τη διατηρήσουμε αλλά και να την αυξήσουμε. με την επίσημη πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας ακόμη και αν λειτουργήσει στην εντέλεια τα τελευταία δέκα χρόνια θα είχαμε καλά αποτελέσματα για τους στόχους της χιλιετίας. Θα είχαμε περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη υγεία. Θα μειώναμε τη δια, τις διακρίσεις ε, κατά των γυναικών. Αλλά θα συνεχίζαμε όμως να, έχουμε, να αντιμετωπίζουμε μπροστά μας ένα βασικό προαναπτυξιακό πρόβλημα αυτών των χωρών. Διότι θα συνεχίζαμε να ενισχύουμε το αποτέλεσμα χωρίς όμως να εξηγαίνουμε τον τομέα τις αιτίες. Δηλαδή τα πραγματικά προβλήματα που θέλουμε να εξομαλύνουμε μέσα από την αναπτυξιακή πολιτική. θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τα αποτελέσματα της ΠΟΕ στην ΤΟΑ. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις φτωχότερες χώρες να, να έχουν περισσότερα εισοδήματα, να τους δώσουμε μεγαλύτερες παραγωγικές δυνατότητες. Όπως είπε ο κύριος Μισελ και όπως σε λίγο θα πει και ο κύριος Γκέρενς, θα πρέπει να διευρύνουμε τη δημοσιονομική μας υποστήριξη διότι όχι απλώς εμείς δίνουμε πόρους αλλά επιτρέπει και υποχρεώνει στην ανάπτυξη δημοσίων διαχειριστικών συστημάτων και όλα αυτά χρειάζονται. Ο κύριος Γκόρη είπε και αυτό είναι ένα σημείο ουσιαστικότατο για την Επιτροπή μας Πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη προπτική. Μια, μια πιο πλευρή εστίαση των δράσεών μας. Αλλά χωρίς να μειώσουμε την δημόσια ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήταν καταστροφικό. Οπότε εγώ συμπέρασμα της τοποθέτησής σας θα έλεγα α συν δέλτα ίσον συν αλλά όχι μείωση. Συμφωνώ με την ιδέα της συνεργασίας νότος-νότος. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε στην ΛΑΧ να αποφύγουμε την ισχύ των, περισσο... των πλέον ηγεμονικών χωρών να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη συνεργασία σε ισότιμα επίπεδα το είδαμε αυτό στη Λατινική Αμερική, δημιουργώντας περιφερειακές, περιφερειακούς θεσμούς με ευρύτερους στόχους πέρα από τη συνεργασία. Κύριε Θεοχάρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και εγώ μέσα στην αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και πραγματικά αναρωτιέμαι αν έχει αλλάξει οτιδήποτε στο στάτους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εξ όσων γνωρίζω θα είμαστε απλώς παρατηρητές. Και αυτό φυσικά μειώνει τις δυνατότητες που έχουμε να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση. Παρακολουθώντας με πολύ προσοχή την ανάλυση, ένιωθα συνέχεια θετικά και αρνητικά συναισθήματα, ζεστό κρύο όπως θα λέγαμε στην Αργό κάποια τελικά συμπεράσματα είναι ότι η ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί είναι πέρα για πέρα πλασματική. Η βοήθεια την οποία προσφέρουμε προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι αναποτελεσματική. Η οποιαδήποτε ανάπτυξη έχει επιτευχθεί, θα συμφωνήσω με τον ε, κύριο Λουί Μισελ, είναι ανισομερής και γι' αυτό δημιουργεί αύξηση και του αριθμού των, ε, των φτωχών παράλληλα με μια αύξηση του πληθυσμού με, όλες τις, ε, συνεπακολουθές, με όλα τα συνεπακολουθά. Συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε την διαφθορά και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι ακριβώς η καλή διακυβέρνηση γιατί αυτό το ζήτημα είναι εντελώ διαφορετικό από τη μια περιοχή στην άλλη. Ε, γι' αυτό το λόγο η, η δικιά μας πρόταση πρέπει να είναι ότι η ανάπτυξη πρέπει να αφορά την κοινότητα ή μικρούς πυρήνες ανάπτυξης, μικρές κυψέλες ανάπτυξης και όχι αυτά τα μαξιμαλιστικά σχέδια τα οποία συνήθως αποτυχάνουν. Η IT το αποδεικνύει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή αυτό που παρατηρείται σήμερα στην IT είναι ανάπτυξη ε, ορισμένων περιοχών ε, ως πυρήνων ανάπτυξης ενώ η γενική εικόνα είναι απογοητευτική αν σε αυτή τη βάση οικοδομήσουμε, νομίζω ότι θα είναι πιο ε, καλή και η παρουσία μας. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις Μαλδίβες και από το πράσινο ακροτήριο. Δεν είναι ούτε ο τουρισμός, ούτε η σεζάρια ευόρα που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην, στο, στην, ε, στο γεγονός ότι δεν ανήκουν πια στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αυτές οι, οι δύο χώρες. Ε, συνεπώς πρέπει να κάνουμε μια πιο καλή αξιολόγηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της κάθε μιας χώρας, να επενδύσουμε πάνω σε αυτά και να παρακάμψουμε ενδεχομένως εκείνα τα οποία δεν γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να μετρήσουμε, δηλαδή την διαφθορά και τις κεντρικές κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Σε ένδειξη αυροφροσύνη προ τον κύριο Κόρ. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα καθυστερημένο. Αυτό όμω που ακούω από πλευρά σα είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ενθαρρυντικά για την Κωνσταντινούπολη. Συμφωνώ πολύ με τα όσα είπε ο κύριο Μισελ μόλι τώρα για την διακυβέρνηση και έχω τέσσερι παρατηρήσει και ερωτήσει ταυτόχρονα. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν, ε, θα πρέπει να ε, επιτελέσουμε το έργο σε κάθε επίπεδο όπως το έχουμε υποσχεθεί. Δεύτερον, ως προς την πολιτική για τα βασικά αγαθά που προτείνεται για την αντιμετωπίση της ε, μεγάλης δεκίμανσης με της πληθυκότητας των τιμών στα βασικά αγαθά. Τρίτον, όταν μιλούμε για διακυβέρνηση, με καταπλήσει το ότι σε αυτά τα πέντε σημεία τη νέα σα αρχιτεκτονική δεν έχετε συμπεριλάβει τη διακυβέρνηση στου πέντε πυλώνε. Και δεν ρωτάμε γιατί. Είναι τόσο ευαίσθητο θέμα η διακυβέρνηση για την UNCTAD και δεν τολμάει να τα εγγίξει. Ε, βλέπει ότι πολλά θα ήταν τα μέλη των ΗΕ που θα θέλουν διαφορετικού χειρισμού και γι' αυτό προτιμά να μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι. Η ανάπτυξη, ξέρετε, έχει να κάνει και με τα κοινωνικά θέματα και με την δικαιοσύνη. Άρα χρειάζεται ένα κράτος το οποίο θα, όχι μόνο θα είναι ισχυρό στις δομές του για να εφαρμόσει πολιτικές, αλλά και θα έχει και το κράτος δικαίου, θα ισχύει το κράτος δικαίου, που θα ορίζει κανόνες τους οποίους, στους οποίους θα πρέπει να υποτάσσονται και οι ταγοί, αλλά χρειάζεται και ένα καλό σύστημα λογοδοσίας. Και εδώ δεν μιλάω για δημοκρατία, μιλάω για λογοδοσία. Αυτό το τρίτο στοιχείο λοιπόν για την εξασφάλιση ενός ισχυρού κράτους, η λογοδοσία, είναι άκρος απαραίτητο και για την αντιμετώπιση της κοινωνικής αδικίας και για να βοηθήσουμε αυτές οι τεράστιες μάζες των ε, κρατών του τρίτου κόσμου να ξεφύγουν από την αθλειότητα στην οποία ζουν. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω ότι διακυβέρνησε αυτούς τους πέντε πυλώνες. Το τρίτο. Τέταρτον, συνοχή οι συνέπειε στις πολιτικέ. Δηλαδή να μην παίρνουμε με το ένα χέρι αυτό που έχουμε δώσει με το άλλο. Το είπατε και εσεί πολύ σωστά. Είναι μια μεταφορική έκφραση την οποία πολύ συχνά χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τι εννοούμε με, τις, με την έννοια συνεπή πολιτική. Αλλά εάν δεν κάνουμε προσπάθεια για τη βελτίωση τη διακυβέρνηση, κατά εμέ τουλάχιστον, γιατί βέβαια ξέρουμε ότι και τα Ε, συμφέροντα του δυτικού και εκβιομηχανισμένου κόσμου δεν πρόκειται να ε, δηλιάσουν μπροστά σε κάποιους ε, τυράννους ή δικτατορίες. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολύ φτωχού ανθρώπους να μην αφήνουμε και ανεξέλεγκτες τις πολύ ισχυρέ και πλούσιες οικογένειες ορισμένων φατριών. Θα πρέπει και εκεί να αναλάβουμε κάποια δράση. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες απόψεις στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Κχετιού, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Εδώ είμαι δίπλα σας, μου βλέπετε. Εδώ είμαι. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την έκθεσή σας εν της ε, διασκέψεως. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν με τόσες εξειδικευμένες γνώσεις συνάδελφοι εδώ. Θα ήθελα μόνο να πω ότι στη τελευταία του σύνοδο το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για τέταρτη διάσκεψη των Παναθηνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες όπου υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα να επικεντρωθούμε κυρίως σε αποτελέσματα και να διατυπώσουμε δείκτες για την μείωση κατά 50% του αριθμού των ΛΑΧ έως το 2020. Ερωτώ λοιπόν εάν θεωρείτε ότι ο στόχος αυτός είναι ρεαλιστικός. Όπως ε, βλέπουμε, δυστυχώς η κατάσταση διαρκώς επιδεινούνται. Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν μεγάλους κλειδονισμούς ε, και χρηματοπιστωτικούς, οικονομικούς καλύτερα και επιστηστική κρίση, βαρθύτατη φτώχεια, ανεργία, διαρθρωτική κρίση. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, η διεθνής κοινότητα δεν έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του προγράμματος των Βρυξελών. Mm. Προγράμματος δράσεως. Δεν έχουμε κανένα δείκτη, λοιπόν, καμιά ένδειξη μάλλον ότι θα πάνε, θα πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα. Και επίση θα ήθελα να υπογραμμίσω και για του συναδέλφου ότι υιοθετούμε κατά τη διάρκεια των ετών πολλά ψηφίσματα όπου όμω ε, δεν προβλέπονται μηχανισμοί επαλήθευση. Και δεν βλέπουμε μηχανισμό που θα μας έπετρεπε για τη συγκεκριμένη περίπτωση να επαληθεύσουμε πώς ή σε ποιο βαθμό έχει υλοποιηθεί το σύνολο των ετοιμάτων του ψηφίσματο. Περιμένουμε από εσά να μα πείτε τι κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου, αλλά εν γέννη ελπίζουμε ότι θα βαρύνουν τρόπον την τα λόγια μα. Πάντω χρειάζεται κάποιο μηχανισμό επαλήθευση. Ε, Πάντω, όπω γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νέε και καθοριστικέ αρμοδιότητε για την έγκριση του αναπτυξιακού προπολογισμού και ελπίζω ότι θα είναι ουσιαστική η επικοινωνία ε, και βέβαια με την έννοια τη λογοδοσία που ανέφερε ο Τάι στον Πέρμα νωρίτερα ε, με το Κοινοβούλιο. Ερωτώ λοιπόν, πώ εξηγείται το γεγονό ότι. Και έτσι έχουμε ουσιαστικά διπλασιάσει την αναπτυξιακή βοήθεια από το 2000 στο 2010 και έχουμε και σημαντικές ενισχύσεις για άμεσες επενδύσεις που επιτρέπουν ε, σημαντική, σημαντική ανάπτυξη σε ορισμένες από αυτές τις χώρες. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, γιατί μένουν τα αναπτυξιακά σχέδια, ε, γιατί υπολείπονται τόσο πολύ των προσδοκιών μας. Έχετε κάποια εξήγηση. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή με τον κύριο Craig Μακέιτ Και θα περιορίσω το χρόνο ομιλία στα πέντε λεπτά, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Θα γνωρίζετε ασφαλώ ότι έχει οθετήσει το Συμβούλιο τα συμπεράσματά του που προσδορίζουν κατευθύνε γραμμέ για τη συμμετοχή στη διάσκεψη τη Κωνσταντινούπολη με βάση και τι συστάσει τη Επιτροπή. Ε, δεν θα τα επαναλάβω, τα γνωρίζετε ασφαλώ πολύ καλά. Δυστυχώ έχασα μεγάλο μέρο τη παρουσίαση του κ. Γκόρ και έχω μελετήσει την έκθεση. κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας ε, για τη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης την προσεχή εβδομάδα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε εν προκειμένου. Η Ευρώπη πάντοτε ε, έδειχνε ενδιαφέρον και προσοχή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της ΛΑΧ ιδιαίτερος και κυρίως αυτές που έχουν προχωρήσει περισσότερο και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός με 53,8 δις ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία, 4,5 δις περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά, με εταιρική ε, σχέση ε, για, τις, ε, για την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας, του 8ου στόχου συγκεκριμένα την εκκριώση της φτώχειας, με εταιρική σχέση για την ανάπτυξη χώρες αυτές και διαφορετικούς ρόλους για τους διάφορους παράγοντες ή θεσμούς που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη για το έγγραφο το οποίο θα προκύψει από τη διάσκεψη της ε, Κωνσταντινούπολης. Οι ΛΑΧ έχουν από πλευρά του όμω και εκείνε ρόλο να διαδραματίσουν σημαντικό και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει και εκείνε να προσδιορίσουν την ε, ε, τις αλλαγές που θέλουν να πραγματοποιηθούν, θέλουν να πραγματοποιήσουν σε συνεργασία με τους εταίρους και χωρικούς. Αυτό είναι ένα αντικείμενο των συστήσεων αυτή τη στιγμή. Έχουμε προσδιορίσει λοιπόν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ότι θέλουμε την ανάπτυξη με βάση του στόχου τη χιλιετία με τρία κυρία θέματα που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε για τη διάσκεψη τη Κωνσταντινούπολης, Όμω τα ξέρετε και σε αυτά τα συμπεράσματα. Πρώτον, καταπολέμηση της, ε, του ευάλωτου χαρακτήρα ε, και τις εκθέσεις του κλειδονισμού των ΛΑΧ, δεύτερον στήριξη μιας ανάπτυξης βιώσιμης και τρίτον ε, στήριξη ανάπτυξης οικονομικής βιώσιμης και διαρκούς στις ΛΑΧ. Δεν νομίζω ότι αυτά έρχονται σε ε, αντίθεση με οτιδήποτε από τα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Εδώ. Όπως είπα, είμαστε ο μεγαλύτερος χωρικός Φυσικά χρειάζεται πολύ περισσότερη βοήθεια για την ανάπτυξη ιδιαίτερα στον ΛΑΧ και θα πρέπει να εξασφαλιστούν και οι κατάλληλε ε, συνθήκε για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Τι ε, δεσμεύσει μα, ε, όχι μόνο για τη χορήγηση βοήθεια, αλλά και με βάση του λοιπού όρου τη πρόταση των Βρυξελών, τη συμφωνία των Βρυξελών, παραδείγματι νεακό αδασμολόγητο, απαλλαγή από ποσοστώσεις κτλ. Τα έχουμε εκτελέσει ως υποχρεώσεις, ε, προχωρούμε ως προς τις απαλλαγές και την ουσιαστική, την ε, ε, ουσιαστική λειτουργία της βοήθειας. Ιδιαίτερα μέτρα για τις ΛΑΧ και τις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν επί παραδείγμα τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλία για την χιλιετία, για την πιστιστική βοήθεια, το Φλέξ. Πρόκειται για δεσμεύσεις που έχει επαναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση 0,7% επί του ΑΕΠ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 0,52% του G8, του ΑΕΠ των G8 για τις ΛΑΧ. Φιλοδοξίες λοιπόν που υπάρχουν και που συνεχίζονται, ενισχύονται και ως προς την πρόσβαση στις αγορές και ως προς άλλα ε, στοιχεία και πολιτικές. Αυτά προς το παρόν. Πιστεύω ότι η συζήτηση σημερινή θα είναι πολύ ε, χρήσιμη και για τη δουλειά μας στην Κωνσταντινούπολη την προσεχή εβδομάδα. Η σε ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γκορ για να διατυπώσει τα συμπεράσματα, να δώσει απαντήσεις του. Και μια και έχουμε καθυστερήσει, παρακαλώ, έστω και με τόσο αυτή συζήτηση, να περιοριστείτε στα 10 λεπτά. Καλώ, λέει ο κύριο Γκόρ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσει. Για να δώσω απαντήσει, σα ξεκινήσω με τι κυρίε, και έτσι επιτρέψτε μου να δώσω απάντηση στις παρατηρήσεις, ερωτήσεις των δύο κυρίων και στη συνέχεια με τη σειρά στους ε, κυρίους. Με συγχωρείτε το όνομά σας, κυρία Θεοχάρους. Είπατε πως σας φάνηκε σαν ψυχρολουσία αυτή η παρουσίαση. Ίσως, ίσως να έχετε δικαιό. Αλλά παρακαλώ μιλήσουμε μόνο ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα και αυτή η τελευταία προγραμματική περίοδος δράση ήταν πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες δύο. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε πιστεύω. Και να έχουμε πάντα υπόψη ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Είναι δυνατόν να αλλάξουν. Μπορούν οι λάχ να τα καταφέρουν. Αυτό. Και δεν θέλω να μείνουμε με την ε, αίσθηση της ψυχολουσίας. Αυτό που θα ήθελα να αφήσω σαν μήνυμα είναι ναι, μπορούν οι ΛΑΧ, ναι, μπορούν και οι αναπτυξιακοί τους εταίροι να τη στηρίξουν στην προσπάθεια αυτή. Η κυρία στα δεξιά μου, λυπούμε και πάλι δεν ξέρω το όνομά σας, η κυρία Γκρέτου, Ρωτάει τι μαθήματα αποκομίζουμε το μεγάλο αυτό, τη μεγάλη αυτή έκρηξη και την κοινωνική ευημερία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ερώτημα και θα πρέπει να το ε, έχουμε πάντα υπόψη. Τι επιδιώκεται τελικά, τι καταφέρνουμε τελικά. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι δεν δόθηκε αρκετή έμφαση στην παραγωγή και την απασχόληση ε, γι' αυτό θα ήθελα να επικεντρωθούμε περισσότερο στην παραγωγή, στη γεωργία, αλλά και εκτός της γεωργίας. Και επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη μεγάλη πρόκληση της απασχόλησης. Τίποτε περισσότερο δεν θα πω προς το παρόν, αλλά πάντως θα ήθελα να επισημάνω ότι θέσετε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και επίσης, η ιδέα αυτή ότι οι, μικρές, οι μισές από τις ΛΑΧ θα έχουν ξεφύγει από αυτό το χαρακτηρισμό σε δέκα χρόνια, στα μισά της περίοδου τέλο πάντων. Είναι για μένα προσωπικά μια φιλοδοξία ίσως υπερβολική. Τεχνικά υπερβολική. Ναι, πλην όμως. Κρίσιμο ερώτημα είναι, πάνω απ' όλα, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει το να έχουμε τις ε, ΛΑΧ που το προτείνουν και οι οποίες λένε θέλουμε εμείς οι, εννιά, μισές από εμά να έχουν ξεφύγει από αυτόν τον ε, χαρακτηρισμό μέχρι το 2020. Νομίζω ότι φιλοσοφικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή όσο προβιβασμός σημαίνει ουσιαστικά ξεφεύγουν από την ε, κατάσταση όπου βρίσκονται σε ένδια και χρειάζονται ειδική διεθνή υποστήριξη. Άρα, όταν μας λένε θέλουμε οι μισές να έχουν ε, προβιβαστεί, ουσιαστικά μας λένε θέλουμε τώρα τη βοήθειά σας για να μην τη χρειαζόμαστε στο μέλλον. Αυτό σημαίνει προβασμός και έχει πολύ μεγάλη σημασία πιστεύω πέραν των τεχνικών δηλαδή χαρακτηριστικών ή στοιχείων. Το 50% των ΛΑΧ ως προοπτική, ως στόχος προβασμού είναι πολύ σημαντικό. Να, θα περάσω τώρα στον Βλή Μισελ, ο οποίος έθεσε ως, ως πρώτη του παρατήρηση αυτό το ζήτημα και αυτό το μύτο της Αριάδνης, της διακυβέρνησης το ζήτημα της διακυβέρνησης που συσχετίστηκε και με την διαφθορά και με το κατά πόσον ε, φέρνει αποτελέσματα η βοήθεια. Ο κύριος Μπέρμαν ρώτησε επίσης γιατί η διακυβέρνηση δεν περιλαμβάνεται στους πυλώνες ε, της διακυβέρνησης. Να σας πω διότι δεν το θεωρήσαμε ως ένα χωριστό κεφάλαιο. Θεωρήσαμε ότι είναι κάτι, είναι ένα στοιχείο το οποίο διαπερνάει, υπάρχει σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι αποφεύγουμε το ζήτημα της διακυβέρνησης. Όχι. Αντιθέτως είχαμε την έκθεσή μας με τίτλο «Διακυβέρνηση, η εξέλιξη στη διακυβέρνηση». Άρα η ανάπτυξη στην διακυβέρνηση, η εξέλιξη μας στη διακυβέρνηση σημαίνει ταυτόχρονα και έκφραση αυτού που θεωρούμε ως έκφραση της καλής διακυβέρνησης. Τι σημαίνει καλή διακυβέρνηση. Έτσι ώστε και όπως είπε και ο Λουί Μισελ να μπορεί κανείς να εξασφαλίσει μια ε, αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό νομίζω αποτελεί στοιχείο της καλής διακυβέρνησης. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει και οι κυβερνήσεις να έχουν μια σαφή ιδέα το πού θέλουν να βαδίσουν, προς τα πού θέλουν να πάνε. Αυτό σημαίνει και καλή επικοινωνία με το λαό βέβαια. Προϋπόθεση για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε να υλοποιήσουμε το όραμα αυτό. έχουμε λοιπόν παραδείγματα, τουλάχιστον πιστεύουμε, ε, κρατών που έχουν καταφέρει σημαντική μείωση της φτώχειας. Και αυτά μας επιτρέπουν να δούμε ουσιαστικά παραδείγματα <laughs> και πάνω σε αυτά μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αναπτύξουν και κέντρα αριστείας στο ιστορικό τους. Οι χώρες αυτές πολλές φορές δεν έχουν ε, τους ε, εγχώριους πόρους. Μερικές φορές δεν είναι καθόλου δυνατόν αυτό. Εάν γιατί είναι 20% του ΑΕΠ ε, που αφιερώνουν οι χώρες αυτές ε, στη διακυβέρνηση. Εάν λοιπόν χάσουν αυτό το 20% μένει πολύ λίγο ποσό. Άρα εξαρτώνται από την εξωτερική βοήθεια. Και όπως επισήμαναν ορισμένοι, όπως και ο Λουί Μισελ, αυτή η σύνδεση, διασύνδεση μεταξύ της διακυβέρνησης και της βοήθειας είναι πολλές φορές τη ρίζα του κακού. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε ίσως να μην ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό και να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα την ιδέα της κυριότητας για τις ίδιες αυτές τις χώρες και να επιτρέψουμε περισσότερο πειραματισμό. Ίσως αυτό βέβαια σημαίνει σημάνει περισσότερες δυσκολίες ως προς τους ε, μηχανισμούς εφαρμογής που έχουμε εδώ η υλοποίηση αλλά θα πρέπει νομίζω να στραφούμε προς την ε, ενίσχυση των ε, ΛΑΧ με βοήθεια, όχι βραχυπρόθεσμη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γίνει τώρα η δραστική αλλαγή. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και χρειάζεται να δώσουμε και ένα περιθώριο για πειραματισμούς στην πολιτική, στη κυβέρνηση. Διάφορα άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Και είναι σημαντικό νομίζω να μην μετατραπεί αυτή η ενίσχυση σε νέα απεικιοκρατία. Αλλά ε, βλέπω ότι υπάρχουν πιθανές και καινοτόμες προσεγγίσεις στην ε, βοήθεια που μπορούν να προκύψουν και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε αυτές τις καινοτόμες προσεγγίσεις, να τις μετατρέψουμε σε βοήθεια. Ο κύριος Γκιουερέρο μίλησε για τεχνολογική ενίσχυση. Βεβαίως και πρόκειται και μία προσέγγιση ε, καινοτόμων που προκύπτει από τις χώρες του Νότου. Επίσης υπογράψε τη σημασία των ε, χωρών του ΠΟΕ. Οι ίδιες οι ΛΑΧ ζητούν πρώιμη συγκομιδή ζητούν ε, δυνατότητες που προκύπτουν από το γύρο της Δόχα να ε, βγουν ουσιαστικά από τα συμπεράσματα της Δόχα προκειμένου να ελοπιθούν νωρίτερα. Ο κύριος Μπέρμαν μίλησε και για τη διακυβέρνηση, ανέφερε όμως και συγκεκριμένα το θέμα της πολιτικής για τις τιμές των βασικών αγαθών. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι ένας διτός στόχος η αντιμετώπιση της πτυτικότητας ή των συνεπειών της πτυτικότητας αυτών των τιμών πρώτον και δεύτερον το να βοηθήσουμε τις λιγότερο εγμένες χώρες να αξιοποιήσουν περισσότερο τους εγχώριους πόρους τους και να διαχειριστούν καλύτερα αυτό το εγχώριο ε, εισόδημα η χρηματοδότηση πιστεύω σε περίπτωση ακραίων συνθήκων θα ήταν ε, μία λύση. Όπως προτείνει η Επιτροπή παραδείγματι ο μηχανισμός FLAX θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα. Επίσης η αξιοποίηση των εγχώριων πόρων θα σήμαινε φερρυπίν την παροχή βοήθειας της ε, ΛΑΧ για μια καλύτερη διάγνωση γεωλογικά του τι είδου σπόρους θέτουν. Οι στόχοι του ΟΝΤΑ θα πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά και θα πρέπει να στραφούμε περισσότερο προς την παραγωγή η, ο τρόπος οργάνωσης των γεωργικών δομών ήταν μάλλον επιβλαβής για τη ΣΛΑΧ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε νέους τρόπους, δημιουργικούς τρόπους, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Ξέρω ότι υπάρχει παρακολούθηση σημαντική από πλευρά σας. Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Πάμε τώρα στα σημεία 6 η εντολή για τον ε, Τρίλογο για το σχέδιο του προπολογισμού του 2012 η Επιτροπή μας προετοιμάζει μία γνωμοδότηση για τον προπολογισμό του 2012. Δέκα λεπτά κύριε Γκέρενς γιατί καθυστερήσαμε. Δεν θα χρειαστώ καν τα έξι λεπτά που μου δώσατε. Πω πω είναι φοβερό να, να, να, να συζητάει κανείς. Διότι σαν να είμαστε στο παζάρι είναι εδώ μέσα και όχι σαν να είμαστε σε συνεδρίαση. Συζητήσαμε ήδη σχετικά. Η Επιτροπή μου ζήτησε να ορίσω καταρχήν τους βασικούς άξονες της Επιτροπής μας, τις βασικές μας προσδοκίες από τον τον επόμενο προϋπολογισμό και εγώ κράτησα καμιά δωδεκαριά σημεία που θα σας υπενθυμίσω. Συμφωνήσαμε στο να ζητήσουμε περισσότερους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από καινοτομή φορολόγηση που θα πρέπει να διερευνήσουμε. αλλά η αρχή μιας νέας και κοινότομης φορολόγησης ε, είναι κάτι το οποίο το συμμερίζεται βρύτατα η Επιτροπή μας. Δεύτερο, στόχοι της ανάπτυξης, κατά πολέμηση της στόχιας καταρχήν. Αν πούμε ότι ο βασικός στόχος είναι η μείωση της φτώχειας, τότε θα πρέπει να δεχθούμε και όλα τα συμπαραμαρτούντα που λένε ότι αν συνεχίσουμε να επενδύουμε σε λάχα, διότι και εκεί πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα σε βάθος. Πριν συνεδριάσουμε εδώ, συναντήθηκα με τους εκπροσώπους της Concord εμείς συζητήσαμε για το κατά πόσο πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την, στην Βραζιλία, στην Κίνα ή στην Ινδία την καταπολέμηση της φτώχειας δεδομένου ότι εκατοντάδες εκατομμυρίων φτωχοί ζουν σε αυτές τις χώρες. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, να προκαλέσουμε αυτές τις χώρες στο να προχωρήσουν σε μία ανακατανομή του πλούτου που δημιουργείται από, την, από το υψηλό αναπτυξιακό τους ποσοστό πολλές φορές πάνω 10%. Αυτοί οι ίδιοι πρέπει να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και όχι ο κοινοτικό προπολογισμό. Η κατανομή του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι από αυτά τα 19 τρισεκατομμύρια των τελευταίων ετών ελάχιστα έχουν κατανεμηθεί, διανεμηθεί στον κόσμο. Τρίτο, για την κλιματική αλλαγή συζητήθηκε στην Κοπεχάγη και θα συζητηθεί και στο μέλλον. Το χρήμα το οποίο επενδύεται για την άμβληση των κλιματολογικών επιπτώσεων στις χώρες αυτές πρέπει να συνεχιστεί. Τέταρτο, τέταρτο, ατόπα, τόπα ήδη. Πρέπει να εστιάσουμε τη βοήθεια στις φτωχότερες χώρες διότι αλλιώς ε, θα διασπαθήσουμε χρήμα στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Πέμπτο. Πρέπει οι λιμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες υπόσχονται πολλά, να μην μείνουν να μην, χωρίς πρικοδότηση. Ας πούμε η, η καταπολέμηση παγκοσμίως ε, της ελονοσίας, της φυματίωσης ε, και του AIDS πρέπει να συνεχιστεί. Ο αρμόδιος επίτροπος με τον αρμόδιο επίτροπο μάλλον το συζητήσαμε στο κοινοβούλιο και αυτός είναι που θα πρέπει να αποφασίσει για την πρόταση για τα κονδύλια. Ξέρουμε όμως ότι πολλές χώρες αντιστέκονται λέγονται, λέγοντας ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε περισσότερο στο, στα κονδύλια για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αλλά η διαχείριση της ενίσχυσης κατά του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας είναι εντελώς άσχετα με όλη την ιστορία της διαφθοράς. Είναι κονδύλια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Επίσης έχω μερικά άλλα για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού και τη συμπληρωματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να πρικοδοτηθεί με ένα κέντρο υποβολής προτάσεων και έρευνας, αναζήτησης καινοτομίας για την ε, αναπτυξιακή πολιτική και βοήθεια και αυτό δηλαδή μετά την συνένωση της Γενικής Διεύθυνσης ε, για την Ανάπτυξη με τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Αυτά προς συζήτηση. Ο κύριος Στάς έχει το λόγο. ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Εξ ονόματος της ομάδας μου Θέλω να σταθώ για, τον για την πρόταση για τον Ευρωπαϊκό Φόρο στον στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τη μείωση της ε, φτώχειας για το θέμα της ε, καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και για τις αναδυόμενες χώρες που θα πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά με βρίσκουν σύμφωνο. Τώρα κάτι άλλο. Εσείς μιλήσατε για τις αλλαγές του κλίματος, αλλά δεν μιλήσατε για περιβάλλον κύριε Γκέρενς. Θα καταθέσω μία τροπολογία αντίστοιχες με τις 44 και 45 της έκθεσης Μίτσελ, επισημένοντας τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και κλίματος και αυτό θα βοηθήσει φυσικά να γίνει σαφέστερη η έκθεσή σας είναι η μόνη μου παρατήρηση ο κύριος Μπέρκμαν ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μερικές παρατηρήσεις αν μου επιτρέπετε καταρχήν η έκθεση του Σάρλ είναι καταπληκτική πρώτο σημείο φόρος στις χρηματοπιστωτικές αλλαγές. Αυτό το ζήτησε το Κοινοβούλιο, πρέπει να προχωρήσουμε. Τα κράτη-μέλη όμως, τα συμπεράσματα τους, ε, του Συμβουλίου μιλάνε για, την, για τις παγκόσμιες συναλλαγές. Αλλά γιατί όμως εμείς εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκό φόρο, γιατί ξέρουμε ότι αν περιμένουμε τον παγκόσμιο φόρο δεν θα, δεν θα δούμε ποτέ προκοπή. Πρέπει να τονίσουμε τη χρηματοδότηση, την ενίσχυση για την καταπολέμηση της στόχιας στις ΛΑΧ. Αλλά με το ICI Plus και το BAM θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί έχουμε, ε, έχουμε πρόβλημα με το Συμβούλιο και την Κομισιόν σχετικά. Πρέπει να αλλάξουμε ίσως τα επιχειρήματά μας γύρω από αυτό. Για τις κλιματικές αλλαγές εμείς οι σοσιαλιστές συμφωνούμε με τον Μπαρτ που λέει ότι και το περιβάλλον θα πρέπει να μπει σε αυτό το σημείο. Μετά, αναδυόμενες οικονομίες, τέταρτο σημείο. Οι περισσότεροι φτωχοί σε αυτόν τον ποταπό κόσμο ζουν ακόμη στην Ινδία, την Κίνα και την Βραζιλία. Και αυτό είναι πλέον διαπίστωση. Και είναι πρόβλημα. Και είναι λάθος να λέμε ότι δεν χρειάζονται αναπτυξιακή βοήθεια αυτές οι χώρες. Νομίζω απλώς ότι χρειάζεται μία βαθμία μείωση αυτής της βοήθειας. Ένα σύστημα συγχρηματοδότησης σε χώρες ε, σαν την Ινδία υπάρχουν ένα σωρό λεφτά για να αγοράζει κανείς τζάγκουαρ ή ε, χαλιβουργίες αλλά δεν έχουν λεφτά για να, προσε... να, να, για να βοηθήσουν τους δικούς τους τους ε, φτωχούς πρέπει να ξεκινήσουμε κοινά σχέδια, να ζητήσουμε συγχρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων. Να σταματήσουμε δηλαδή αυτήν την... Ε, ε, να, να, να φτάσουμε μάλλον στην απεξάρτηση ε, της χώρας από τη βοήθεια. Για την αναπτυξιακή βοήθεια και το 10% εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια τρύπα στο νερό. Κύριε Γκέρενς, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ορίζουμε ποσοστά. Θεωρούμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα είναι όλο ένα και, θα, είναι όλο ένα και πιο απαραίτητη στο μέλλον. Διότι και με την, με, με την αστιφιλία κάθε θεομηνία όλο ένα και περισσότερες ζημιές προκαλεί και περισσότερα θύματα έχουμε. Χρειάζεται λοιπόν, ε, θα, θα μας στοιχίζει πολύ πιο ακριβά όλα αυτά. Χρειάζεται κάτι να κάνουμε, δεν θα χάνουμε μόνο ανθρώπους, θα χάνουμε και κτίρια. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οργανωτικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ Θα επιμείνω στη θέση ότι σε καμία χώρα η οποία αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και επενδύει σε ε, διαστημικά προγράμματα δεν πρέπει να δίνεται αναπτυξιακή βοήθεια, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα των πυρηνικών όπλων. Γι' αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε ε, κάθετοι. Έχουν αρκετά λεφτά για να κάνουν ό,τι κάνουν με τα πυρηνικά, ας τα διαθέσουν για τον κόσμο. Τώρα, ένα ειδικό θέμα είναι αυτό που έχει πει ο κύριος Γκέρνς και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά χαίρομαι που είναι κοινή διαπίστωση ότι θέματα υγείας που αφορούν την καταπολέμηση του AIDS, της ε, φυματίωσης, της ελονοσίας, τη χάνουν ειδικού χειρισμού και διατίθενται σημαντικά κονδύλια και χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε και κάποιε άλλε νόσου, αυτέ τι νόσου των φτωχών όπω λέμε ή τι νόσους που θα μπορούσαν να θεραπευτούν με απλά θεραπευτικά σχήματα ή τι γαστρεντερίτιδε που αποτελούν μια σημαντική αιτία θανάτου παιδιών ε, ειδικά στον τρίτο κόσμο και με απλά μέσα όπω με τη διάθεση χνοστοιχείων ψευδαργύρου νέων φαρμάκων τα οποία έχουν ανακαλυφθεί μπορούμε να ρυθμίσουμε, να αναστείλουμε μάλλον την θανατηφόρο δράση αυτών των ασθενειών. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό τομέα στον οποίο πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να ε, διαθέσουμε περισσότερα κονδύλια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Thank you, Madam Chair. And, uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. ευχαριστώ του κυρίε και κύριου βουλευτέ για τι παρατηρήσει σχετικέ με τον προπολογισμό. Πρόκειται για μια στιγμή όπου όντω καλούμεθα να αναλογιστούμε τις διάφορες ε, αιτίε των περικοπών ή τη στενότητα των πόρων στο τμήμα 4, στην κατηγορία 4. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αναλογικότητα μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι η ανθρωπιστική βοήθεια ενδεχομένω υποχρηματοδοτείται αλλά και ότι κάθε ανθρωπιστική αλλά και ανθρωπιστική, ε, αναπτυξιακή αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια στο παρελθόν ήταν υποχρηματοδοτημένες. Από την άλλη, ανθρωπιστική βοήθεια ίσως δεν είναι ε, αυτή η οποία επιτρέπει την εγγραφή ενός συγκεκριμένου ποσοστού γιατί οι ανάγκες από έτος σε έτος μπορεί να ποικίλουν και άρα ε, πρέπει η εγγραφή συγκεκριμένων ποσοστών επί του προϋπολογισμού να αναφέρεται περισσότερο σε αναπτυξιακή βοήθεια. Ίσως λοιπόν μπορεί μακροπρόθεσμα ως προς τις ε, αιτήσει να είμαστε κάπως πιο δίσκαμπτοι αλλά από την άλλη έχουμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις ως προς τις δαπάνες σε αναπτυξιακή βοήθεια. Για τα διάφορα άλλα θέματα που επισημάνθηκαν. Με ενδιαφέρον άκουσα τα σχόλια για την Ινδία και την Κίνα, τη Βραζιλία. Ξέρω ότι είναι ακαθόδης ε, χώρος. Είναι θέματα τα οποία έχουμε επισημάνει και στην Πράσινη Βίβλο. Και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε μια ανακοίνωση για τις ε, συνέπειες αναπτυξιακής πολιτικής, όπου θα εξετάζουμε τα διάφορα θέματα της Πράσινης Βίβλου και θα διατυπώνουμε συγκεκριμένες προτάσεις από αυτών. Οι προτάσεις πιστεύω θα δώσουν απαντήσεις σε κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την πρόσβαση στην ιδιωτική ε, χρηματοδότηση, στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Ε, είναι ένα ζήτημα, το γνωρίζουμε, πρόβλημα στον χώρο της αναπτυξιακής βοήθειας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και ως προς το ζήτημα των ε, συνεπειών της αναπτυξιακής βοήθειας. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπε ο κ. Μισελ νωρίτερα. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέπει να καταδεικνύουμε τα επιτεύγματα και τον απόϊχο της αναπτυξιακής μας βοήθειας. Εν τέλει θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερος ότι συζητούμε ένα νέο οργανικό γύρο διαπραγματεύσεων στην ΤΕΦΚΟ και ίσως έτσι μπορούμε να δώσουμε απάντηση και στις ανησυχίες του κυρίου Γκέρενς για την πολιτική, την αναπτυξιακή και τη, και τη νέα ε, διατύπωσή της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Σύντομα παρακαλώ για να καταλήξει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται προκάλεσα πολλούς όταν είπα ότι δεν χρειάζονται οι χώρες αυτές ε, δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Η συζήτηση συνεχίζεται και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Μου αρέσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι συνάδελφοι διάβασαν προσεκτικά την έκθεση, ιδίως εδώ μπροστινός μου. Ακόμη και αν διαφωνούμε, είναι κάτι πολύ θετικό το γεγονός ότι τουλάχιστον διάβασε αυτά που έγραψα. Εδώ θα είμαι πολύ, θα επιμείνω πολύ. Υπάρχει ανέχεια και μέσα στην Ένωση, την οποία δεν έχουμε καταπολεμήσει επαρκώς χρησιμοποιώντας τα ταμεία της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας. Το ίδιο ισχύει και για τις αναδυόμενες χώρες που έχουν πόρους και θα ήθελα να μου εξηγήσει η Κομισιόν γιατί να συνεχίσουμε να τιμωρούμε τα προγράμματα που να μην τιμωρούμε προγράμματα που δεν διαθέτουν τα χρήματα που έχουμε εμείς προβλέψει ως βοήθεια. Η κυρία Θεοχάρου με υποστήριξε από αυτού και την ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει απόλυτα δίκιο. Εδώ είναι ευθύνη των αναδειωμένων χωρών των ιδίων. Άλλο θέμα, η σχέση ανθρωπιστικής με αναπτυξιακή βοήθεια. Πάντοτε βέβαια πρέπει να προέρχονται τα ποσά από τα αρμόδια ταμεία, αλλά αν θέλουμε να διαχωρίσουμε την ανθρωπιστική από την αναπτυξιακή βοήθεια και τη συνεργασία, θα βλέπαμε ότι η πρώτη, η ανθρωπιστική δηλαδή, συνήθως ανταποκρίνεται σε κάποια αποτυχία ενώ η δεύτερη είναι επένδυση προς το μέλλον. Έχω και εγώ κάποια πολιτική εμπειρία και ξέρω ότι 10% για την ανθρωπιστική και 90% για την αναπτυξιακή θα μου φαίνονταν καλή ιδέα. Έπειτα δεν άκουσα κανέναν να διαφωνεί με αυτά που έγραψα για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών δοσοληψιών. Το σημειώνω αυτό και επανέρχομαι στην προβληματική των αναδειωμένων. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας απότομης παύσης της βοήθειας. Θα ήθελα όμως προοδευτικά να αντικατασταθούν οι δωρεές της Ένωσης από εισφορές των ίδιων των χωρών. Ε, αφού συμφωνούμε τόσο το καλύτερο. Μπορούμε να καταλήξουν τα πράγματα όμορφα. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 5 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, σημείο 7 συζήτηση των 68 τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο έκθεσης του κυρίου Γκέρενς για το μέλλον του της αναπτυξιακής βοήθειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχετε πάλι το λόγο κύριε Κιόνης για αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω από την αρχή ότι δεν έχω σκοπό να συζητήσω και τις 68 τροπολογίες. Δεν θέλω καν να το κάνω. Θέλω απλώς να σας πω τι περίπου είναι το πνεύμα τους. Γενικά και οι 68 τροπολογίες κινούνται μεταξύ ευφορίας και αμφιβολιών. Δηλαδή, είτε υπερτιμούν ε, τη βοήθεια που μπορούμε να χορηγήσουμε, είτε είναι ζητούν υπερβολικά μεγάλη δημοσιονομική φρόνηση. Συγκεκριμένα θα ήθελα να κάνουμε το εξής. Δεν είμαι σίγουρος για πολλές τροπολογίες γιατί το μείγμα τόλμης και φρόνησης δεν είναι πάντοτε το σωστό. Αν απορρίψουμε μερικές τροπολογίες στις οποίες ο συντάκτης επιμένει για υπερβολική φρόνηση στη χρήση του προϋπολογισμού δεν θα έχει άδικο μεν. Αν όμως αυτό είναι το μόνο του επιχείρημα τότε αυτό για μένα είναι προβληματικό. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε ορισμένους κινδύνους. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τη δουλειά μας αποκλείοντας κάθε κίνδυνο. Η συνεργασία για την ανάπτυξη υλοποιείται μέσα σε ένα πολύ μετάβλητο πλαίσιο και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στην έκφραση που λέει ότι καλύτερα να βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία ως μισογεμάτο ποτήρι παρά ως μισοάδιο. Το περιεχόμενο του ποτηριού είναι πάντοτε το ίδιο, είτε το βλέπουμε ως μισοάδιο είτε ως μισογεμάτο, αλλά το θέμα είναι αν η τάση του είναι προς το γέμισμα ή όχι. Άρα πρέπει να δούμε τα πράγματα αλλιώς από το αν το μισό ποτήρι σημείωνε την τάση να αδειάσει παραπάνω. Δεν είναι το ίδιο. Αν η δυναμική είναι δυναμική βελτίωσης λοιπόν, δεν είναι το ίδιο με το αν είχαμε μια δυναμική χειροτέρευσης. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή που πρέπει να εκτελέσει αυτά τα προγράμματα, η Κομισιόν, να εκτιμήσει ποιος ακριβώς είναι ο αναλήψιμος κίνδυνος. Οι περισσότερες τροπολογίες λοιπόν είτε εφορία, χαρακτηρίζονται είτε από εφορία είτε από σκεπτικισμό και αμφιβολία. Εγώ θα έλεγα ότι για την αναπτυξιακή συνεργασία από τον περασμένο αιώνα έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που μπορούμε να τα ε, περιγράψουμε ως εξής. Πρώτα η αποαπικιοποίηση, μετά η βοήθεια η οποία συνεχίστηκε, εφαρμόστηκε με τρόπο μάλλον πατερναλιστικό. Επόμενη, στην επόμενη φάση απαγορευόταν να τίθενται όροι. Η Κομισιόν σταμάτησε αυτή την πρακτική την οποία θεωρούσα και εγώ ανεύθυνη γιατί δικαίω θεώρησε ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι όροι ή έγινε μια κίνηση αποκεντρωτική και μέσα σε αυτή τη λογική χορηγείται και η βοήθεια που χορηγείται σήμερα. Βέβαια πρέπει να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, η διαχείριση, ο έλεγχος. Η διαχείριση του κινδύνου όμως δεν μπορεί να αποφευχθεί με την αρχή όμως της αναλογικότητας. Έχω σοβαρές ανησυχίες ως προς, το, ως προς αυτά που συμβαίνουν σήμερα για το Ταμείο Καταπολέμησης του AIDS, της Ελλονοσίας και της φυματίωσης. Έχει υπάρξει κάποια κατάχρηση ποσών και αυτό είναι σκανδαλώδες Αλλά δεν πρέπει αυτό να οθήσει τους δωρητάς να πάψουν τη χορήγηση της βοήθειας. Ορισμένοι το κάνουν για το 2011 τουλάχιστον. Αν συνεχίσουν αυτήν τους τη στάση, τότε αυτό που θα γίνει μάλλον είναι ότι θα πληρώσουν την ύφη οι ασθενείς και οι πτωχότεροι. Πρέπει εδώ να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέτρα. Έπειτα Ορισμένες τροπολογίες πρέπει να δούμε, να μας πει η Κομισιόν μάλλον ποιες τροπολογίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσκολία στη διαχείριση του προϋπολογισμού αυτού. Αν υπάρχουν τροπολογίες που αμφισβητούν τη δυνατότητα αυτή από την Κομισιόν να μας το πει. Αν δεν αντιτίθενται δηλαδή στην ίδια τη λειτουργία και εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκέρεντς. Το συζητήσαμε σε, μια, παλιότερη συνεδρίαση της Επιτροπής και τότε είπα ότι και εγώ ήμουν ένα ημισηγητής ε, για το ίδιο θέμα στα πλαίσια της ΑΚΕ, της αντιπροσωπείας ΑΚΕ. Και προβλέψαμε να συναντηθούμε σε δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη. Και σε παλιότερες συνεδριάσεις της ΑΚΕ, για να συνεχίσω το σκεπτικό του κυρίου Γκέρελτς, διαπιστώσαμε ότι οι θέσεις ε, πάνε στα δυο άκρα. Την άκρα τη εφορία από τη μια και τον σκεπτικισμό, τον άκρατο σκεπτικισμό από την άλλη. Την απόλυτη αποδοχή με την απόλυτη απόρριψη. Είναι λοιπόν καιρός στις πολιτικές συνεργασίες να αναλάβουμε ρίσκα και να κάνουμε και αλλαγές. Εγώ εντάσσομαι στην ομάδα των τολμηρών. Όχι βέβαια των α, ε, κατεχομένων από εφορία, αλλά τέλος πάντων α, ε, μεταξύ των α, ε, αισιοδόξων. Καλύτερος όρος από την εφορία ή τον ενθουσιασμό. Με, τον όρο όμως του να δίνεται λογαριασμός. Δηλαδή να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν, πώς χρησιμοποιούνται στο μέλλον όλα αυτά, πώς λειτουργούν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ότι δεν λειτουργεί σωστά ή να ενισχύσουμε αυτό το οποίο λειτουργεί. 11 τροπολογίες κατέθεσα, το ένα έκτο δηλαδή συνολικά των τροπολογιών του κυρίου Γκέρεντς. Και αυτές οι, οι τροπολογίες στείνουν στην κατεύθυνση της ελεγχόμενης τόλμης. Ζητούνε να υπάρχει μία διαβάθμιση. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε και μετά να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και με κεντρικό ρόλο σε αυτό το μέσο. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικό, πρέπει να είναι συμβατό με άλλους τρόπους βοήθειας. Θα πρέπει να αποφύγουμε τους όρους. Δεν θα ήταν συμβατό με τον προϋπολογισμό. Πρέπει να βρούμε κίνητρα, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός να καταπολεμάει τη φτώχεια, ορισμένες ασθένειες, να βοηθάει στην εκπαίδευση, στην υγεία κλπ. Και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημοσιονομική ενίσχυση για να ενισχύσουμε τον δημόσιο τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες, την governance, την εύνομη διακυβέρνηση και διαχείριση. Και οι χώρες δικαιούχοι της βοήθειας να μπορούν να υπόκεινται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των κοινοβουλίων τους. Να ενισχύσουμε τις ικανότητες, τις διακυβερνητικές ικανότητες των κυβερνήσεων αυτών των χωρών και ο έλεγχος να γίνεται από την δική τους κοινωνία των πολιτών, τα δικά τους κοινοβούλια. Ευχαριστώ ο κύριος Στάς. Καθυστερήσαμε να είστε σύντομος. παίρνω το λόγο μέσα από έναν διπλό ρόλο. Εισηγητής στον έλεγχο του προϋπολογισμού και μέλος της Επιτροπής. Και ξέροντας τι γίνεται στην Κοκομπή, δηλαδή τολμηροί και σκεπτικιστές, στην Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού και εκεί στη μάχη, τη μάχη φαίνεται την κερδίζουν οι σκεπτικιστές. Πάντως αυτή η έκθεση χαρακτηρίζεται από ισορροπία, δηλαδή τολμηρή χρηματοδότηση αφενός, αλλά αφετέρου πρόβλεψη ορισμένων ελέγχων και φραγμών. Εγώ με τον ε, συνεισηγητή έχω, με τον εισηγητή συγγνώμη, έχω υπογράψει 13 ε, τροπολογίες και εμεί το 1 τρίτο δηλαδή οι τροπολογίες 40 και 42 λένε ότι θέλουμε να αυξήσουμε την ε, αυτονομία των χωρών δικαιούχων και σε άλλες συζητήσεις και σε άλλες εκθέσεις είναι ένα σημείο το οποίο επικαλούμε θα τακτικά. Θέλουμε επίσης αυτές οι χώρες να προετοιμάσουν με τα κοινοβούλια τους στρατηγικές οι οποίες δεν θα είναι κάθετες όπως προτείνει η Κομισιόν. Θα πρέπει και τα τοπικά κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχουν και αυτά τη γνώμη τους. Η τροπολογία 59 είναι σημαντική για μας. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη συζήτηση. Πρέπει εμείς να ενισχύουμε χώρες οι οποίες έχουν επαρκή ε, ορυκτό πλούτο και πετρέλαιο. Πρόκειται για το facing out το οποίο ζητάμε και για τις τροπολογίες 21 και 22 λέμε ότι η δημοσιονομική βοήθεια θα πρέπει πάντα να αποτελεί μια προσωρινή μεταβατική λύση μέχρι τη στιγμή που αυτές οι χώρες δικαιούχοι της βοήθειας θα μπορούν μοναχές τους να διαχειριστούν την κατάσταση και θα έχουν και ένα φορολογικό σύστημα που θα τους επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτούνται. Αυτός θα είναι και ο ίστατος στόχος μας. Ο κύριος Κέσλερ. Ευχαριστώ πολύ. Και ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω εκ μέρου του ΕΡΚ τον κύριο Γκέρεν για τη δουλειά του. Μερικά πράγματα τα επεξεργαστήκαμε από κοινού στι ε, τροπολογίε. Και θα ήθελα προκαταβολικά να διατυπώσω μια επικριτική ίσως παρατήρηση προς τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι με καταπλήσει το γεγονός ότι το monitoring και η αξιολόγηση ε, από ό,τι φαίνεται ξεφεύγουν από την έννοια του ελέγχου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τους συναδέλφους από την Επιτροπή των Προπολογισμών και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να διεκδικήσουμε αυτή τη ε, διάσταση. Και επίση, όπω λέει ο κύριο Γκέρεν, ταυτόχρονα βλέπουμε ότι έχει ε, πραγματοποιηθεί ένα θέμα προ την ορθή κατεύθυνση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη και για κίνητρα στο πλαίσιο του προπολογισμού, δηλαδή δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και ομολογόμενο ότι εγώ από την εμπειρία που έχω, έχω μάλλον επικριτική στάση ως προς την ενίσχυση μέσω του προπολογισμού, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί να ζητούμε περισσότερα για τα περισσότερα χρήματα που δίνουμε και περισσότερα αποτελέσματα, more for more, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο σωστός δρόμος και επίση, νομίζω ότι θα πρέπει στην αρχή και την έννοια του capacity building να εισαχθούν, να αναπτυχθούν νέε ιδέε για το τι μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και ω εκ τούτου κατέθεσα και τι σχετικέ τροπολογίε, τι προσωπικέ μου τροπολογίε, την ιδέα του της φορολογίας DVTX 2020, 2020 πώς δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά να ε, διαμορφώσουν τις ε, δημοσιονομικές τους δομές κατά τρόπον ώστε να είναι βιώσιμες και μέσα από αυτή την ε, ε, ενίσχυση από τον προπολογισμό να τους βοηθήσουμε να στηριχθούν πάνω σε δομές αξιόπιστες και ουσιαστικές. Αυτά θα ήταν κάποια κίνητρα τα οποία πιστεύω μπορούμε από κοινού να ε, ενισχύσουμε. Αποφεύγοντας ταυτόχρονα και κάποιες αρνητικές εκδηλώσεις ή αρνητικά στοιχεία τα οποία έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Νικολέτα Μέρλο από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν χαίρεται ιδιαίτερα για την υποστήριξη της Επιτροπής σας έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της στήριξης προϋπολογισμών και θα συνεχίσει να αποτελεί αυτό σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή συνεργασία και στο μέλλον. Έχουν Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότητά του και γι' αυτό θα συνεχίσουμε την εφαρμογή του μέσου αυτού. Θα ήθελα να σας δείξω σε ποιους ακριβώς τομείς η πολιτική αυτή έχει φέρει αποτελέσματα. είναι προβλε... υπάρχει μεγάλη προβλεψιμότητα και γι' αυτό παραμένουμε δεσμευμένοι σε μια πολιτική που μπορεί να μετρηθεί, να έχει αυτά αποτελέσματα. Όποτε βέβαια υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Θέλουμε με βάση αυτή την εμπειρία να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των χωρών που θέλουμε να βοηθήσουμε. Δεύτερον, συμφωνούμε με την Επιτροπή σας ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν διαδικασίες ε, που να διασφαλίζουν ότι θα είναι υπόλογοι οι χρήστες για την χρήση και θα είναι πιο μεγάλη η συμμετοχή όλων των παραγόντων στην εφαρμογή των προγραμμάτων <clears throat> έτσι ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα των σωμάτων και οργανισμών αυτών στις τρίτες χώρες για αυτολειτουργία. Σύμφωνα βέβαια όλα αυτά με τις συστάσεις της τελευταίας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Η σύσταση 20 δείχνει ότι προσπάθειά μας για καλύτερη στήριξη πρέπει να γίνει ακόμη πιο μετρήσιμη και αποτελεσματική. Αλλά βέβαια δεν λέει τίποτα για την κακή χρήση ή κατάχρηση. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη μείωση της ανέχειας, αλλά επίσης για να υπάρξει μεγαλύτερο αίσθημα του ανήκειν στις κοινωνίες αυτές. Όλα αυτά για μας είναι πολύ σημαντικά και τα λαμβάνουμε υπόψη και στα κριτήρια επιλεξιμότητας των προγραμμάτων αλλά και στους διαλόγους συνεννόησης ανάλογα με το, την κάθε χώρα βέβαια. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπουμε κάθε φορά ποια είναι η πραγματική κατάσταση της κάθε χώρας, όπως λέει και η σύσταση 51. Σε σχετικά πλουσιότερες χώρες, τα προγράμματα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια για την χρήση των φυσικών τους πόρων. Επίσης, η στήριξη αυτή δεν είναι το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη. Υπάρχουν και άλλα. Ε, ευχαριστώ παιδί μου αρκεί. Λοιπόν θα δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. είπα τα ουσιαστικά στην εισαγωγή μου. Προτείνω μία μέθοδο για να ολοκληρώνουμε. Προτείνω να συνεδριάσουμε με τον κύριο Στάντος γύρω από να βρεθούμε και να συμφωνήσουμε γύρω από το συμβιβασμός και να δούμε και με την Κομισιόν ποιες από τις τροπολογίες θα είναι οι πιο ενοχλητικές σε ορισμένες από τις τροπολογίες. Αν θεωρείτε ότι ορισμένες τροπολογίες καθιστούν την πολιτική μη λειτουργική θα πρέπει να το επιχειρηματολογήσετε. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. και εμπλούτησαν τις συζητήσεις μας με τη συνεισφορά τους που είναι σημαντικότατη. Να σας ε, τιμήσω ότι στις 25 Μαΐου τελειώνει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Ψηφίζουμε γνωμοδότηση της Ισαμπέλ Λεβίν. Έχετε όλη την κάρτα ψηφοφορίας να κάνουμε μία δοκιμή. Να βάλετε την κάρτα σας στην σχετική υποδοχή για να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Α, μάλιστα. Εγώ ψήφισα ναι, ναι, ναι. Έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα, πρέπει να τελειώνουμε πριν από τα μεσάνυχτα λοιπόν. Il y a 22 votants, c'est... Voilà, c'est bon, d'accord. Oui. Ah oui. Donc on peut voter. Can we vote in block? I don't know what the other groups are, but I only have... Να ψηφίσουμε en block, Δεν ξέρω τι λένε οι άλλες ομάδες. Μα και εγώ αυτό ήθελα να σας προτείνω. Αν δεν έχετε πρόβλημα, βεβαίως. Ψηφίζουμε. Α, κάποιος δεν συμφωνεί. Τροπολογία 1. Διανατάσεως της χειρός. Mm. κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οι τέσσερα καταπίπτει. Πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. αν δεν είναι εδώ η συγγήτρια. τώρα Πάμε τώρα. Στη γνωμοδότηση του κυρίου Σβένσον. Τροπολογία 1. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά θες να να ελέγξεις, ναι, ναι, θα το ελέγξουμε. Τη 2, ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Ρεστε 3. Απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία της Γιουδίθ ε, Σαρτζεντίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7. Κυρία Πρόεδρε, δεν πέρασε η ένα. Οπότε έχει καταπέσει αυτή η τροπολογία. Σωστά, σωστά, σωστά. Η έξι έχει καταπέσει. Ψηφίζουμε την 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οχτώ. Οχτώ. Υπέρ. Κατά. Κισαψτιά. Αποχές. Αμάντμαν νεφ. Εννιά. Oui, αμάντμαν, Εννιά είπα. Υπέρ ατά, χες μα δεν ψηφίζει κανείς θα επαναλάβουμε 9 δεν ψηφίσατε λοιπόν με τις κάρτες άρχεται η ψηφοφορία την τροπολογία 9 ψήφισαν όλοι και όλες έλειψη ψηφοφορία εγκρίνεται Δέκα υπέρ κατά χες απορρίπτεται. Έντεκα υπέρ κατά από χες εγκρίνεται. Δώδεκα υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Δεκατρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε όλες μαζί μέχρι και την 21 μάλιστα Η γραμματεία μου λέει ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός εδώ και αν γίνει δεκτός ο συμβιβασμός θα καταπέσουν οι υπόλοιπες. Λοιπόν, χωριστά, 18 υπέρ. Κατά, χες, εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Υπέρ της συμβιβαστικής. Κατά συμβιβαστικής. Αποχές εγκρίνεται. Άρα μέχρι και την 21 κατά Την 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Πε. Τα. Χες. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα υπέρ κατά χες απορρίπτεται 28 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 29 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 30 σε τμήματα πρώτο τμήμα είπα 30 χωριστά. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Πώς καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Μάλιστα τότε ηλεκτρονικά το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξαν, δεν ψήφισαν όλοι, ούτε όλες. Λείπει ένας ή μία. Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ ομοφωνία δηλαδή. Τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Μίτσελ. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 έχει καταπέσει. Τροπολογία 14 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Τα χες εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. χες απορρίπτεται. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ. Κατά. χες εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ 17 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 18 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 19 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 Προφορική τροποποίηση, μάλιστα. Α, υπάρχει νέα μορφή του. Α, η τροπολογία 21, αλλά με προφορική προφορική τροποποίηση. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 22 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, Τροπολογία 21 λέει ο Πρόεδρος υπέρ. Είχαμε δεχτεί την προφορική και τώρα τη γραπτή. Λοιπόν, υπέρ της 21, κατά της 21, αποχές απορρίπτεται. Τώρα 22 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 πώς όχι θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 22. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έληξε. Εγκρίνεται Τροπολογία 23 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Δε, ε, κατά. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική. Πρώτο τμήμα της 23. Άρχεται η ψηφοφορία. έληξε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 34 υπέρ τα χες απορρίπτεται 35 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 36 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 περ κατά αποχές εγκρίνεται 40 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση μάλιστα για την 44 ηλεκτρονική επαλήθευση αρχή τέλος εγκρίνεται 45 υπέρ α χες εγκρίνεται έχουμε μια δυσκολία. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. χες εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. χες εγκρίνεται. Μετά έχουμε μια προφορική τροπολογία των πρασίνων σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εδώ υπάρχει κάποια σύγχυση. Γιατί είχε προβλεφθεί μία ψηφοφορία και τώρα γίνονται δύο. Εγώ νόμιζα ότι θα γινόταν μία ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία, αλλά τώρα είναι σε δύο τμήματα. Ναι. Δεύτερο τμήμα λοιπόν της 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. έντεκα υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Το υπόλοιπο του σκεπτικού. Όλα τα υπόλοιπα. μέχρι το 6 όλα μαζί υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται το 6 καταπίπτει και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφοφορία έληξε εγκρίνεται ομόφωνα Δεν υπάρχουν διάφορα δυστυχώς. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας γίνεται στα Σβρυξέλλας την 3η 24 Μαΐου 3 με 6.30 και την Τετάρτη 25 9 με 12.30 και 15 με 18.30. Θα συνεχίσουμε εδώ μέσα τη συνεδρίαση των συντονιστών και συντονιστριών και παρακαλώ όσους δεν είναι συντονιστέ και συντονίστρια να φύγουν από την αίθουσα, να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Oui, je la salle. Ça va.